Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ καθίστε. Gestern keine Zeit gefunden. Äh, Χτες δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε τη συζήτηση ε, για την έκθεση της κυρίας Λόζεν και ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη. Προτείνουμε τώρα λοιπόν πριν την ψηφοφορία να γίνει η συζήτηση. Σύντομα να μας παρουσιάσει η κυρία Λόζεν την έκθεσή της. Αν θέλουν να μιλήσουν και οι σκιώδεις εισηγητές, καλώς. Και μετά να πάμε στην ψηφοφορία για να συμπεριλάβουμε όλα αυτά που θα έχουμε ακούσει την ψηφοφορία μας. Η έκθεση είναι της Επιτροπής Ανάπτυξης, με εισηγητή τον κύριο Ντέβα, η δική μας είναι γνωμοδότηση. Έχετε το λόγο λοιπόν κυρία Λέζεν. Ευχαριστώ πολύ, θα είμαι σύντομη κι εγώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για την πολύ καλή συνεργασία και ιδιαίτερα τους συναδέλφους. Ήταν πολλές επικοδομητικές οι ε, προτάσεις τους και οι τροπολογίες. Συμφωνούμε όλοι και είμαστε πεπισμένοι ότι η αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να έχει στόχο την καταπολέμηση της ένδυας και την εκρίζωσή της. Και συμφωνούμε επίσης όλοι ότι ο στόχος που έχει σημασία είναι η βοήθεια να φτάνει εκεί που χρειάζεται, στον τελικό της αποδέκτη. Φυσικά, πρωταρχικός στόχος είναι αυτός. Και βέβαια οι ιδιωτικέ εταιρείε δεν έχουν ως στόχο να αναπτύξουν τις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται, αλλά στόχος τους είναι η κερδοφορία. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, τεκμηριωμένα στοιχεία που λέγουν ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κανόνες. Η αρπαγή γεών, το περίφημο land grabbing στην Αφρική, οργιάζει. Γι' αυτό ζητούμε δεσμευτικές προδιαγραφές διεθνείς και υποχρεωτικές για τις εταιρείες. Ε, υπάρχουν ευρωπαϊκές εταιρείες που οθούν εκτός της αγοράς ε, τις ντόπιε εταιρείε αυτών των χωρών, πράγμα που εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Στόχος λοιπόν της νομοδότησης είναι να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς οι ιδιωτικές εταιρείε μπορούν να βοηθήσουν για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλές ήταν οι τροπολογίες οι οποίες ε, είχαν να κάνουν με τις ευκαιρίες και με τα όρια ε, των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη. Ε, καταλήξαμε σε κάποιους συμβιβασμούς και ελπίζω οι συμβιβασμοί στους οποίους καταλήξαμε να βρουν πλειοψηφία στην ψηφοφορία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριο Πλένκοβιτς. Αξιότιμη κυρία Λόζινγκ. Ο κύριος Κιουτσούκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι στις τροπολογίες φαίνεται η σημασία του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να πετύχουμε τους βασικούς στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της φτώχειας. Θέλουμε να οδηγηθούμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και όντως μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλει αλλά βέβαια μπορεί αυτό μόνο να γίνει αν παράλληλα προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αν προωθούμε επίσης ε, το κράτος δικαίου και τον ε, εκδημοκρατισμό. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα συγκεκριμένες ρήτες ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί τμήμα όλων των νέων συμφωνιών που θα υπογράφουμε στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα περίοδο προγραμματισμού. Σα καλώ λοιπόν να υποστηρίξετε τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιτσούκ. Ο Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ. Ε, ο σκιώδη εισηγητής μας, ...κύριο Στετίνα, απουσιάζει για να σας διηγηθεί τι τράβηξε στο διάλογο ε, για αυτή τη γνωμοδότηση, η ομάδα μας αποφάσισε να την καταψηφίσει, διότι παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν, ε, έχει ιδεολογική φόρτιση. Μαρξιστική, λενινιστική ε. θεώρηση για τον ιδιωτικό τομέα είναι η γνωμοδότηση αυτή και δεν μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε ε, ιδεολογικές τοποθετήσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Ο κύριος Χάουιτ, παρακαλώ. Ρίτσαρτ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της ομάδας ε, πρέπει να πω ότι θα υπερψηφίσουμε τη γνωμοδότηση παρότι γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι του ΕΛΚ ε, έχουν επιφυλάξεις. Στη συνεδρίαση των σκιωδών είδα ένα κείμενο που έχει περισσότερο σχέση με το πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο παρά με το θέμα. Ε, Κάποιο έλεγε ότι ο ειδικό τομέα δεν έχει ρόλο στην ανάπτυξη και μια άλλη ομάδα έλεγε ότι είναι ε, οι πρωταθλητές και θα πρέπει αυτού να προωθούμε και κανέναν άλλον. Εγώ εξ ονόματο της ομάδας μου είπα και λέω κάτι πιο λογικό, ότι έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει ο ιδιωτικό τομέα και το ε, αναγνωρίζουμε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική εταιρική ευθύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό το θέμα τη αρπαγής των γεών έχει σημασία και ζητούμε περισσότερα από τους ιδιώτες και θα ήταν κρίμα να μην περάσει αυτή η γνωμοδότηση ε, από ανθρώπους που δεν ξέρουν πολλά πράγματα για το θέμα. Εγώ είμαι αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχω γνωρίσει επιχειρηματίες που δείχνουν πολύ περισσότερη ηγετική στάση από ό,τι καμιά φορά εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να παίρνουμε το καλό παράδειγμα ίσως από αυτούς. Ευχαριστώ ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το που είπε ο συνάδελφο του ΕΛΚ. Θεωρούμε τη γνωμοδότηση αυτή βασικά ιδεολογικά ορμόμενη από την άκρα αριστερά και θα την καταψηφίσουμε. Ο κύριο Σαφχάουζερ, παρακαλώ. Ε, ναι, πρόεδρε. Η έκθεση... Η έκθεση αυτή έχει θετικά στοιχεία, πρέπει να το αναγνωρίσουμε ας πούμε. Δείχνει πόση φοροαποφυγή, το βάρος, το άχθος του χρέους που είναι ένας από τους κύριους λόγους έλλειψης ανάπτυξης της Αφρικής. Αλλά, ε, αλλά και εγώ είμαι ικανοποιημένο από την υποστήριξη για τις μικρές επιχειρήσεις, την στήριξη του ιδιωτικού τομέα και για την ανάπτυξη και η έκθεση αυτή έχει ένα κρατιστικό όραμα και προσέγγιση που έχει αποτύχει στην Αφρική. Στην Αλγερία ας πούμε ή σε άλλες χώρες που προσπάθησαν να εφαρμόσουν τέτοια μαρξιστικά πράγματα βρέθηκαν τελικά σε πολύ δύσκολη κατάσταση έλλειψης ανάπτυξης ακόμα χειρότερα και από τις άλλες χώρες. Θα καταψηφίσουμε λοιπόν αυτή την έκθεση παρά ορισμένα θετικά στοιχεία που έχει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαφχάουζερ. Κυρία Λούζινγκ, euh, έχετε να πείτε τίποτα πριν την ψηφοφορία σας παρακαλώ. Τι να πω τώρα εγώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισσότερα. Ε, με ξανά και ξανά ότι σε πολλά θέματα δεν συζητούμε επί της ουσίας, αλλά με αιτιάσεις και κατηγορίες τις οποίες αποκρούω. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήταν πάρα πολύ ισορροπημένη η προσέγγιση στη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση και μπορούμε να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Πάγιο. Ces amendements. Λοιπόν, ψηφίζουμε κύριε μου και κύριοι. Συμβαστική 1. Θεέ μου τώρα μπλέκουμε. Τμήμα πρώτον. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο. Dagegen. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο θέλετε, καλώς. 24 υπέρ 35 κατά, με μικρή διαφορά απορρίπτεται, λέει ο Πρόεδρος. Τι είναι αυτό τώρα που δεν μπορώ να διαβάσω εδώ. Μα είναι λαμπουρνέζικα αυτά που μου γράφετε εδώ geschrieben. Was soll der Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, στην τροπολογία 1. Όχι, καταπίπτει λέει εδώ. Αν εγκριθεί η συμβαστική. Και πάμε στην 8 λοιπόν. Wer ist für Antrag 8? Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. Η τροπολογία 10. Υπέρ. Ε, κατά. απόχέ εγκρίνεται. Η 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. wurde Α, η 8 απερίφθη. Λάθος έκανα τότε. Ε, ψηφίζουμε τότε την 11, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 35 υπέρ, 21 κατά. 3 συμβαστική, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 τροπολογία τώρα. Υπέρ κατά αποχές απορρίφτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική 5 τώρα λοιπόν υπέρ. Κατά Enthaltung. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 56. Μποργέζιο είπε. Κατά. Αποχές απορρίψετε. 57 είπε, Κατά. Αποχές απορρίψετε. 59 είπε, Κατά. Αποχές απορρίψετε. Συμβαστική 6 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όλα τα υπόλοιπα πέφτουν 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 79 τώρα. Υπέρ Κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ αρχίζει. Die Abstimmung ist geschlossen. Εγκρίνεται 34 υπέρ 30 κατά. Ε, κυρία Λόζινγκ. Κυρία Λόζινγκ, παρακαλώ. Η ομάδα μου στην τελική ψηφοφορία υπερψήφισε τη γνωμοδότηση αυτή διότι θέλουμε με όλους τους συμβιβασμούς να εγκριθεί και να προχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχουν θέσεις σημαντικές για μας ε, που δεν εγκρίθηκαν. Αποσύρω το όνομά μου από τη γνωμοδότηση αυτή. Dann wird es ein namenloser Bericht. Τότε θα είναι ανώνυμη έκθεση, η γνωμοδότηση. Διότι ούτε ο πρόεδρος θέλει να συνδέσει το όνομά του με αυτή τη γνωμοδότηση. Herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Wir kommen jetzt zum Thema Libanon. Πού πάμε τώρα στο Λίβανο. Ματίας εδώ η κυρία Ματίας. Πάμε λοιπόν στο σημείο 10. Ενημέρωση σχετικά με τη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση στη Βηρητό. Ήταν η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες μας ΡΕΚ. Η κυρία Ματίας ήταν η κυρία Μανέσκου εκεί, ο κύριος Κοσολίνο και η κυρία Βίνμπερχ. Αυτή ήταν η αντιπροσωπεία μας Βηρητό. Έχετε το λόγο κυρία Ματίας. Περιμένουμε λιγάκι. Παρακαλώ σταματήστε τις ιδιωτικές συζητήσεις σας για τα πηγαδάκια. Εκεί οι σοσιαλιστές είναι δύο με μαλλιά εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και η αντιπροσωπεία που είχε πάει στο Λίβανο 16 με 20 Ιουνίου, μόλις επέστρεψε δηλαδή, αποτελούνταν από τέσσερις ευρωβουλευτές εμένα ως προεδρεύουσα αντιπρόεδρος ήταν η κυρία Μανέσκο και Κρίστιν και Ανδρέα Κοσολίνο. Η αποστολή λοιπόν αυτή α, δεν μ' ακούει ο πρόεδρο τέλο πάντων μιλάω και δεν μ' ακούνε. Τέλος πάντων η αποστολή αυτή ήταν σημαντική, αλλά έγινε ακόμη πιο σημαντική μέσα στη συγκυρία που ζούμε. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όπως και στη Συρία έτσι και στο Λίβανο. Φυσικά αυτά οφείλονται στον πόλεμο στη Συρία και θα ήθελα να καταλήξω σε ορισμένα συμπεράσματα από την επίσκεψη αυτή. Εσείς τα μέλη λάβατε την ανακοίνωση τύπου που προετοιμάσαμε στο τέλος της ε, αποστολής και τα κύρια συμπεράσματα ήδη εμφανίζονται εκεί. Πρέπει να τα έχετε δει. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι όσο συντομότερη γίνεται. Ήθελα λοιπόν να πω απλώς τα εξής για το περιεχόμενο της επίσκεψης. Και μετά θα κάνω και ορισμένες αναλυτικές και πολιτικές παρατηρήσεις. Το περιεχόμενο λοιπόν της επίσκεψης. Δύο μέρες αφιερώσαμε για την κατάσταση στο Λίβανο και μία ημέρα στην κατάσταση στη Συρία. Για την κατάσταση στη Συρία. Όταν φτάσαμε στο Λίβανο συναντήσαμε εκπροσώπους των αρχών όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και τον Πρωθυπουργό τον Πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπους τεσσάρων πολιτικών ομάδων κομμάτων δηλαδή για, δηλαδή το κίνημα μέλλον, το Χεσμπουλά τον κ. Ανάναούν, και τον εκπρόσωπο του Ναμπίγ Δεν μπορέσαμε όμως να συναντήσουμε τον Τσαμπίν Ζαζά ούτε τον Βαλίτ Τζουμπλάτ για λόγους ανηλυμένων υποχρεώσεων. Είχαμε προβλέψει συναντήσεις. Και εκτός αυτού συναντήσαμε και εξέχοντα μέλη του στρατού μη κυβερνητικέ οργανώσεις και εκπροσώπους οργανισμών του ΟΗΕ που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Θα ήθελα απλώ να πω τρία πράγματα. Πρώτον, κάτι για τη γενικότερη κατάσταση στο Λίβανο, δεύτερον για την κρίση των προσφύγων και τρίτον για τη Συρία. Συρία. Η Κριστίνα Βινμπέργκ είναι παρούσα, δεν ξέρω αν είναι και οι άλλοι εδώ. Μανέσκου και Κονσολίνου δηλαδή, θα ζητήσω από τη συνάδελφο Χριστίνα να προσθέσει αν θέλει κάτι σε αυτά που θα πω. Για το Λίβανο λοιπόν. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την υπάρχουσα πολιτική κατάσταση και προφανώς, αυτό μου φαίνεται εμένα προφανές δηλαδή, ο ρόλος μας ήταν να ενθαρρύνουμε τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στο Λίβανο να ξεπεράσουν το θεσμικό αδιέξοδο για να υπάρξει εγγύηση καλής λειτουργίας των εθνικών θεσμών. Ιδιαίτερα θίξαμε το θέμα των προεδρικών εκλογών και συμμεριζόμαστε όλοι την άποψη ότι e ότι οι ίδιες οι αρχές του Λιβάνου πρέπει να αποφασίζουν για την τύχη τους και όχι εμείς. Μιλήσαμε λοιπόν γι' αυτό γιατί ήταν ουσιώδες. Τώρα, για τους Σύρους πρόσφυγες. Το 2013 προείδρευσα μιας άλλης αποστολής στο Λίβανο και τότε ο αριθμός των σύρων προσφύγων ήταν ήδη 300.000. Εκείνη την εποχή λέγαμε ότι είχε είχαν ξεπεραστεί τα όρια. Η χώρα έχει 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόνο και τον πληθυσμό που ξέρετε και υπάρχουν Παλαιστίνοι και Σύροι πρόσφυγες Δύο εκατομμύρια περίπου προσφύγων δέχεται ο Λίβανος, στο Λίβανο. Είναι πολύ βαρύ για μια τόσο μικρή χώρα. Ένας στους τρεις κατοίκους του Λιβάνου είναι πρόσφυξ. Και αυτό σημαίνει ότι, ότι λέγω, ότι αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες αλληλεγγύης του Λιβανέζικου λαού αναγνωρίζουμε τον βασικό ρόλο που παίζουν ε, οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και η αποστολή μας, η αντιπροσωπεία μας προσπάθησε να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος που βεβαίως είναι κατεπήγον αλλά δεν αρκεί μια τέτοια προσπάθεια, είναι προφανές. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο όμως πρέπει να τηρήσει στεναρή στάση ως προς την ευρωπαϊκή ανταπόκριση για την υποδοχή των προσφύγων. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι έσχος η κατάσταση αυτή. Και και το ότι μερικές χώρες αρνούνται να δεχτούν μερικές εκατοντάδες προσφύγων ενώ χώρες σαν το Λίβανο φέρουν το βάρος 1,5 εκατομμυρίου σύρων προσφύγων αυτή τη στιγμή. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία επίσης να επισκεφθούμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να δούμε ένα προσωρινό στρατόπεδο κατασκήνωση προσφύγων όπου είδαμε οικογένειες που ζούσαν εκεί. Δεν μπορούν να συνεχίσουν τα πράγματα έτσι. Ένα στα τέσσερα παιδιά μόνο πηγαίνει στο σχολείο. Ο ΙΕ και η πάτη αρμοστία του για τους πρόσφυγες μπόρεσαν να μοιράσουν, να δώσουν μόνο 19 δολάρια αναπρόσφυγα. Κάτι πολύ λίγο δηλαδή. Θυμάμαι ότι κάθε οικογέ... συριακή οικογένεια για να μπορέσει να μείνει σε, ένα... μια προσωρινή κατασκήνωση, καταβουλισμό, χρειάζεται 50 περίπου δολάρια το μήνα και 50 δολάρια το μήνα η εκπαίδευση. Όταν λοιπόν ο ΙΕ δεν έχει να δώσει παρά μόνο 19 δολάρια το μήνα αναπρόσφυγα, αναγεγραμμένο πρόσφυγα, αυτό σημαίνει ένα τεράστιο βάρος όχι μόνο για τους ενδιαφερόμενους αλλά και για την κοινωνία του Λιβάνου, για τις οικογένειες του Λιβάνου οι οποίες επιδεικνύουν τεράστια αλληλεγγύη υπάρχουν όμως όρια και σωματικά και υλικά όρια και γι' αυτό οι αρχές του Λιβάνου προσπάθησαν να κλείσουν τα σύνορα τα έκλεισαν μάλλον και δεν δέχονται πλέον άλλους πρόσφυγες. Είναι όμως ζωτικό το πρόβλημα, κρίσιμη η κατάσταση. Ο ΙΕ και ορισμένοι εμπειρογνώμονες του που συναντήσαμε μας λένε ότι δεν είναι ρεαλιστική λύση αυτά τα προσωρινά μέτρα διότι ο Λίβανος περιτριγυρίζεται από το Ισραήλ, τη Συρία και τη Μεσόγειο. η δε κατάσταση στη Συρία έχει επιπτώσεις πάνω στο Λίβανο φυσικά. Ήδη στην ανακοίνωση τύπου μας το λέμε ότι λαμβάνοντα υπόψη μας όλες τις προσπάθειες αλληλεγγύης που κάνουν οι Λιβανέζικες και οι οικογένειες και οι αρχές και ο λαός ολόκληρος, λαμβάνοντα υπόψη τις τεράστιες χρηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ επιτόπου, επίσης δεδομένων όλων όσων σας είπα, πρέπει να γίνει μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την Ένωση από την Ένωση λέγω για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση να μην κάνουμε στουρθοκαμιλισμούς αφού μας λένε ότι λείπουν χρήματα εγώ δεν ήμουν παρούσα όταν μιλούσε η κυρία Μογκερίνη αλλά χθε διάβασα τις αποφάσεις που ελήφθησαν 12 εκατομμύρια ευρώ έχουν προβλεφθεί Νομίζω με τα 12 αυτά εκατομμύρια μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά είναι θέμα βέβαια πολιτικής επιλογής. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ποια πολιτική επιλογή θέλουμε να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και πώς θα κατανείμουμε αυτά τα χρήματα των φορολογουμένων καλύτερα. Τα 12 εκατομμύρια λοιπόν για τις, για τις περιπόλους είναι κάτι που δεν θα λύσει το πρόβλημα βέβαια των προσφύγων. Θα μπορούσα να πω καλά περισσότερα. Καταφέραμε να αφιερώσουμε μία μέρα στην κατάσταση, για την κατάσταση στη Συρία. Συναντήσαμε πολλούς πρέσβεις της Ένωσης και πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους. Συναντήσαμε την κυρία Κουαλαμάτα που είναι τμήματάρχης ματάρχης λέγω του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Συρία και μπορέσαμε να πάρουμε άμεσες πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Δυστυχώς δεν πήγαμε στη Συρία αλλά, αλλά αυτό θα συζητεί. Τι? E και άλλη φορά. Πρέπει να σας μεθυμίσω ότι το προσδόκιμο ζωής στη Συρία από το 11 έχει περάσει από τα 75 στα 55 χρόνια. 20 χρόνια χάθηκαν από προσδόκιμο ζωής τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Αυτό λέει πολλά. Είναι ουσιώδες, αυτό ήθελα να σας το τονίσω. Και κάτι άλλο που μας το είπαν επιτόπου και εκπρόσωποι του ΟΗΕ και πρέσβης και άλλες αντιπροσωπείες. Okay, ε, και... Τι μας είπανε λοιπόν, τι μας είπανε, μας είπανε ότι, μας είπανε ότι τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης, ναι, τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης, τα κυριότερα μέσα ενημέρωσης λένε ότι μεταξύ Νταές και Αλνοστρά υπάρχει διαφορά. Η μία οργάνωση είναι πιο ριζοσπαστική από την άλλη, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μετριοπαθείς τρομοκράτες. Ο καθένας βέβαια χρησιμοποιεί τις εκφράσεις που θέλει, αλλά πάντως οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε σε αυτές τις διαφοροποιήσεις μεταξύ τρομοκρατών. Υπάρχει τρομοκρατική απειλή τόσο από τον ΤΑΕΣ όσο και από το Αλνούσαρα και η έκκληση της κυρίας Μάτα ήταν σαφής να αποφεύγουμε τέτοιες διαφοροποιήσεις η προσπάθειά μας πρέπει να είναι συλλογική, κοινή, ώστε η καταπολέμηση της τρομοκρατίας να μπορεί να είναι αποτελεσματική. Να μην διαχωρίζουμε λοιπόν πράγματα που δεν είναι χωριστά και που δεν τα βλέπουν ούτε οι επιτόπου άνθρωποι. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό και σχετικό με αυτό που είπα είναι η έκκληση των κατοίκων Δηλαδή τα όπλα των τρομοκρατών. Πρέπει να σταματήσουμε τέτοιες δοσοληψίες ώστε αυτοί που εκπαιδεύουν τους τρομοκράτες για να πολεμήσουν στη Συρία να εμποδιστούν. Αλλιώς ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και επιτρέπουμε τη συνέχιση των σφαγών και όχι το σταμάτημά τους. Με τη χρηματοδότηση λοιπόν την πώληση όπλων σε τρομοκράτας είτε τους θεωρούμε σε εισαγωγικά είτε όχι και όπως σας είπα αυτό δεν ισχύει και δεν το βλέπουν ούτε κάτι και εκεί όταν λοιπόν πολλούνται όπλα σε τρομοκράτας συνεχίζουμε να είμαστε συνένοχοι των τρομοκρατών. Πριν από την επίσκεψη αυτή είχα ήδη πιστεί ότι υπάρχει ανάγκη να οργανωθεί η επίσκεψη και άλλες επισκέψεις στη Συρία και τώρα είμαι ακόμα πιο πεπισμένη. Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα, σαν να μην έχει σχέσεις με τη Συρία το Κοινοβούλιο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επισκεφτούμε τη Συρία ως αντιπροσωπεία και να κάνουμε επαφές με την κυβέρνηση, με το καθεστώς, με τις αρχές και το τοπικό κοινοβούλιο αλλά να γίνει αυτή η προσπάθεια. Επαναλαμβάνω να γίνει επίσκεψη χωρίς αμαλγάματα και συγχύσεις. Ξέρουμε ότι έχουν διακοπεί οι σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά να γίνει η επίσκεψη. χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτού του ταξιδιού και την αντιπροσωπεία, ιδιαίτερα τη Μαρίσα Ματίας, η οποία ηγήθηκε με πάρα πολύ υποδειγματικό τρόπο σε μια αποστολή και αντιπροσωπεία με πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη αυτή η αντιπροσωπεία και πραγματικά είδαμε διάφορα πράγματα που μας γέμισαν με φρίκι. Είχαμε επαφές ε, με κυβερνητικές ε, πλευρές, με πολιτικά κόμματα, μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις. Ήταν τόσο πολλές εντυπώσεις που αποκομίσαμε και μεταφέραμε που θα χρειαστούμε χρόνο για να τις επεξεργαστούμε, για να τις χωνέψουμε. Μας είπε ένας βουλευτής ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα ο Λίβανος. Και επίσης μας είπαν ότι υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα δημόσιας υγείας. Έτσι και πάθεις καρκίνο στο Λίβανο, χάθηκες. Εκατομμύρια, ε, πάνω από ένα εκατομμύριο οι πρόσφυγες δεν έχουν υδροδότηση, δεν έχουν ηλεκτροδότηση. Είναι πραγματική κρίση τεράστια και ο κόσμος χρειάζεται βοήθεια. Ο λαός του Λιβάνου κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη βοήθεια. Ε, δεν αρκούν τα μέσα που διαθέτουν. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να γίνει. Και δεν μόνο αυτό. Ε, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχουν κατακλειστεί από τόσο κόσμο. Είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο να ενταχθούν, βρίσκονται σε σύγκρουση και ανταγωνίζονται και διαγωνίζονται για τις λίγες θέσει εργασίας. Το ένα πρόβλημα οδηγεί στο άλλο, ενός μύρια έπονται, ένα στα τέσσερα παιδιά πηγαίνει σχολείο. Μα είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση. Δεν μπορείτε καν να το διανοηθείτε αυτό που συμβαίνει εκεί. Σε καταβλισμό προσφυγικό ένα παιδί, ένας έφηβος 13-14 χρονών που δεν ε, πηγαίνει σχολείο είναι πολύ ε, εύκολο να πέσει στα χέρια των ε, τρομοκρατών και να στρατολογηθεί. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση, σχολεία, βοήθεια. Ο ΦΑΟ βοηθάει βέβαια στη Συρία ε, και στο Λίβανο, ε, αλλά χρειάζεται και εκεί η βοήθεια. Ε, χρειάζεται μια ελπίδα και ένα μέλλον να τους δώσουμε, να τους υποσχεθούμε. Τι άλλο να πω. Το σημαντικότερο, το είπαν και οι περισσότεροι, ήταν αυτή η ροή προσφύγων, η κρίση και η αγωνία και ο φόβος της τρομοκρατίας. Ε, αυτό το είδαμε παντού από όλους τους συνομιλητές σχεδόν που μας το έθεσαν υπόψη. Και όπως είπε και η Μαρίζα, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να στείλουμε αντιπροσωπεία και στη Συρία την ίδια, για να δούμε ε, εκ του σύνεγγυς τα πράγματα. Δηλαδή το να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε είναι πολύ εύκολο, αν δεν έχεις ιδέα τι κατάσταση επικρατεί επί τόπου. Ούτε εγώ έχω συγκεκριμένη λύση για τα προβλήματα αυτά. Ε, δεν μπορούμε παρά να ευχηθούμε ειρήνη και στη Συρία και παντού σε όλο τον κόσμο. Ε, εύκολα είναι να τα λες αυτά. Το δύσκολο είναι να κάνεις αυτό που χρειάζεται. Ε, χρειάζονται πηγόντως βοήθεια αυτοί οι άνθρωποι, τρόφιμα, τα βασικά, δυνατότητες εκπαίδευση και περισσότερα κονδύλια αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντιπροσωπή αυτή. Με βοήθησε πάρα πολύ, έμαθα πολλά πράγματα και τα σημειώνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δεν έχω πολλά πράγματα να προσθέσω σε αυτά που ήδη υπόθηκαν από τις συναδέλφους μου που πήγανε μαζί μου στο Λίβανο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι μας έκανε εντύπωση όλες εκείνες τις μέρες και έχει να κάνει με τους καταβλισμούς προσφύγων. 1.200 μόνο και μόνο στο Λίβανο. 1.400.000 Σύριοι, 800.000 στην Τουρκία, εκατοντάδες χιλιάδες στην Ιορδανία. Αυτό που κάνει λοιπόν εντύπωση είναι οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτούς τους καταβλισμούς προσφύγων. Οι περισσότεροι είναι νέοι ως 18 ετών και οι άνθρωποι αυτοί από ιδεολογικής πλευράς, κοινωνικής πλευράς δέχονται πιέσεις συνεχώς από τις τρομοκρατικές οργανώσεις και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πώς θα καταφέρουμε να βρούμε πόρους και κονδύλια για να πετύχουμε μια πολιτική ισορροπία στο Λίβανο. Η χώρα αυτή έχει παραλύσει πολιτικά. Ήρθαμε σε επαφή με τον Πρωθυπουργό και ακόμα και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για τον επόμενο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων που θα διοριστεί σύντομα στη χώρα αυτή. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους καταβλισμούς προσφύγων. Πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως εκεί τελικά νεκραγούν τα πράγματα, ιδίως όσον αφορά την επιρροή που ασκούν στους νέους οι α, τρομοκρατικές οργανώσεις. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της πολιτικής γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένω να πρέπει να μας δοθεί μια κάποια νέα αρμοδιότητα για να τα αποκριθούμε και στους νέους αυτούς τις χώρες αυτές. Να καταφέρουμε δηλαδή να προωθήσουμε περισσότερο και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους νέους αυτούς για να μην χάσουμε όλη αυτή τη νέα γενιά, για να μην χάσουμε τους νέους και κυρίως τα παιδιά. Να προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε μια διεθνή διάσκεψη με βασική πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με συνεργασία άλλων διεθνών φορέων προκειμένου πραγματικά να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε με τους νέους στους προσφυγικούς καταφλισμούς. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους. Έχουμε αρκετούς σπόρους, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να τους διοχετεύσουμε περισσότερο προς πιο συγκεκριμένους στόχους. Να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους μας για να βοηθήσουμε τους, νο... τους νέους αυτούς. Θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε καλύτερα και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το μέλλον της όλης αυτής περιοχής. Όσον αφορά τη Συρία, μας έκανε προφανώς εντύπωση οι ε, επαφέ που είχαμε την Παρασκευή το πρωί με του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στη χώρα αυτή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει τελικά με την πόλη του Αλέπο και του του Χαλεπιού τις επόμενες εβδομάδες πολλά πράγματα διακυβεύονται εκεί πέρα. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τη Συρία. Ας προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε τελικά να επανακαταστήσουμε εκεί πέρα έναν διάλογο κυρίως με το Κοινοβούλιο της χώρας, το Κοινοβούλιο της Συρίας. Κυρία Λιωμαρή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη της αντιπροσωπείας για την έκθεσή τους είναι πάρα πολύ εύγλωτη και υπογραμμίζει τα διάφορα στοιχεία της κατάστασης των σύρων προσφύγων εκεί. Υπάρχει ένα σημείο που νομίζω δεν αναπτύχθηκε πάρα πολύ και θα με ενδιέφερε και μου είχαν επιστήσει την προσοχή σε ένα ταξίδι που είχα πάει πέρσι στο Λίβανο και έκτοτε συνάντησα ξανά Λιβανέζους φίλους μου είναι πώς επηρεάζει τη ζωή του Λιβάνου και την ισορροπία του Λιβάνου αυτή η ροή προσφύγων. Διότι πέρα από τα θεσμικά προβλήματα Υπάρχει ένα βασικό θέμα εκεί, ας πούμε, πώς ε, επηρεάζει ε, την εργασία των Λιβανέζων. Έχουν μεγάλο ανταγωνισμό, είναι πολύ πιο μικρή αμοιβή που δίνεται στους πρόσφυγες. Επίσης, ε, στη στέγη έχουν αυξηθεί τα ενίκια, γιατί έρχονται Σύριοι που έχουν χρήματα και έρχονται να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά της στέγης. Ε, ε, ε, μου λένε ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Επίσης, στα πολιτιστικά και στην ισορροπία. Σύριοι και Λιβανέζοι δεν ταυτίζονται ακριβώς ως προς την κουλτούρα και ε, τα χαρακτηριστικά τους. Ε, και ε, το ίδιο ισχύει για την Ιορδανία. Το είπε και η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου που πήγε στην Ιορδανία. Αντίστοιχα, πολύ σημαντικά. Το ταμείο που αναφέρατε είναι σημαντικό ως ιδέα, διότι θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος ενδεχομένως λοιπόν από τους Σύρους πρόσφυγες σε όλη την περιοχή και η Ευρώπη δεν έχει πόρου, είναι τελείως ανεπαρκής. Από την άλλη, αν ε, δημιουργηθεί ένα ταμείο, θα μπορούμε εκεί να συνδυάσουμε πόρου που προέρχονται από άλλε χώρε τη περιοχή, βλέπε χώρε Περσικού κόλπου και κάποιε άλλε, που ε, ενέχονται πάρα πολύ ε, και ενδιαφέρονται να υπάρχει ασφάλεια στο Λίβανο, στην Ιορδανία και γενικότερα στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν συζητήθηκαν αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, αν σας τα έθεσαν υπόψη συνομιλητές. Ο κύριο Κόουσο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία ε, και θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Όταν συναντηθήκατε με την εκπρόσωπο του κυρίου Δημιστούρα, όταν ήρθε εδώ μας είπε ότι εργάζεται για να υπάρξουν εστίες κατάπαυσης του πυρός. Τι γίνεται, έχει γίνει αυτό, ε, για να, ε, θα βοηθούσε πάρα πολύ τον πληθυσμό που τόσο πολύ έχει υποφέρει. Ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Συριακή κυβέρνηση και τις επισκέψεις. Εγώ είμαι υπέρ. Όχι μόνο να πάμε, να συζητάμε και με την κυβέρνηση. Γιατί όχι, με όλους πρέπει να συζητάμε. Πρέπει να έχουμε όλους τους διάβλους επικοινωνίας ανοιχτούς προς όλους. Δεν είναι σαν τράπηδες όπως η Σαουδική Αραβία που περιφρονεί τις γυναίκες, αποκεφαλίζει και διώκει πολιτικά κόμματα. Αν δεν είναι δικός μας. Δηλαδή. Και είναι και ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους μάλιστα παρόλο που χρηματοδοτούν αυτού του τρομοκράτε, έχουμε τι πιο αγαστέ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία. Τρομοκράτε που στη συνέχεια έρχονται και επιτίθεται στην Ευρώπη. Ε, όχι μόνο υποστηρίζω να πάμε στη Συρία αλλά να μιλήσουμε με όλου όσοι ενέχονται στη σύραξη γιατί είναι ο μόνο τρόπο να λυθεί. Ευχαριστώ πολύ. <coughs> Ε, Μίκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω πάει στη Συρία, τέσσερις μέρες ε, ήμουν εκεί. Συζήτησα με διαφόρους, με ανθρώπους τους οποίους εσείς δεν μιλάτε. Και ε, τι έχει σημασία κατά την άποψή μου, να αναλύσουμε την κατάσταση πιο πολύ από το να πάμε, τη στρατιωτική κατάσταση δηλαδή. Η μόνη δυνατότητα να αποφευθεί ολοκαύτωμα με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς είναι να υποστηρίξουμε την εξοχότητά του τον Μπασάρα Λάσατ. Είναι η μόνη πιθανότητα και δυνατότητα να αποφύγουμε καταστροφή. Μπορεί να σας αρέσει, να μην σας αρέσει ο κύριος Άσατ, αλλά πρέπει να καταλάβετε το εξής. Ο δημοκρατικός στρατός έχει όπλα που πάνε στο χαλιφάτο μετά από τρεις μέρες. Ναι, ναι. Λέτε νέα διάσκεψη. Ωραία, νέα διάσκεψη πρέπει να βοηθήσουμε το μόνο άνθρωπο που μπορεί να έχει μια διαφορετική Συρία. Ούτε Σουνίτες, ούτε Σιήτες, ούτε Χριστιανούς, ούτε τίποτα. Μια Συρία ε, πολυπολιτισμική. Αυτός είναι η εξοχότης του ο Μπασάρ Ελ Άσετς και θα πρέπει ε, να αποταθούμε σε αυτό τώρα, γιατί μετά από ένα εξάμεινο θα είναι κατόπιν εορτής. Ευχαριστώ πολύ. Τι είπε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω τι ακούσαμε για αυτό το τελευταίο θέμα. Μάλιστα το μέλλον της Συρίας πρέπει να καθοριστεί από τους ίδιους τους κατοίκους της. Πρέπει όμως να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν τα πάντα που χρειάζονται ώστε να μπορέσει ο λαός της Συρίας να πάρει μόνος του τις αποφάσεις του. Η πολιτική λύση που θα βρεθεί δηλαδή για την ε, κρίση στη Συρία πρέπει πρώτα να τη φανταστούμε. Τώρα για τη δυνατότητα οργάνωσης τρίτης διάσκεψης αναφερόσασταν σε κάποια Γενέβη 3 ή κάτι τέτοιο. Δεν είμαι βέβαιη ότι το κατάλαβα καλά. Δεν μπορούμε να περάσουμε σε Γενέβη 3 αν δεν κλείσει πρώτα πλήρως η διαδικασία Γενέβη 2. Πρέπει να μπορέσουμε δηλαδή να ασχοληθούμε να κλείσουμε πρώτα την, την προηγούμενη διάσκεψη πριν προβλέψουμε επόμενη και να βρεθούν πολιτικές και ειρηνικές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιοχή. Για το πρώτο θέμα η κατάσταση στο Λίβανο και οι επιπτώσεις της, στη ζωή των ανθρώπων εκεί. Ναι, το είπαμε διαμακρού. Μιλήσαμε και για θέματα κοινωνικού dumping, αυξανόμενη ανεργία, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στο Λίβανο. Η ανεργία έχει αυξηθεί. Και όταν μιλήσαμε με πρόσφυγες από τη Συρία μας είπαν ότι μπορεί να υπάρχει παιδί που μαζεύει 25 κιλά παλιοσίδερα την ημέρα και κάτι ανάλογο ισχύει και για γυναίκες που πληρώνονται πριν πολύ λίγο δυσαναλόγως σε σχέση με την προσπάθεια που κάνουν και υπάρχει παιδική εργασία διότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο ακούσαμε αυτά που μας είπαν και, και οι δύο άλλοι συνάδελφοι πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια αγγίση ότι θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο τα παιδιά μόνο ένα στα τέσσερα πηγαίνει τα υπόλοιπα δουλεύουν για ένα δολάριο την ημέρα. Είναι λοιπόν σημαντικό το θέμα κοινωνικά, όχι μόνο το κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά και άλλα θέματα στέγαση, είδωρ, ηλεκτρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, όλα αυτά. Και νομίζω λοιπόν ότι Έχουμε πολλή δουλειά. 10.000 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι μόνο ο Λίβανος. Ας πούμε, εφαρμόστε κάτι ανάλογο στην Πορτογαλία. Αν μεταφέρουμε την πραγματικότητα εκεί θα σήμαινε ότι η Πορτογαλία πρέπει να δεχτεί 20 εκατομμύρια πρόσφυγες κάντε το και εσείς υπολογίστε με τις χώρες σας. Ανάλογα με τον πληθυσμό της Πορτογαλίας που έχει 10 εκατομμύρια θα είχαμε 5 εκατομμύρια αν το υπολογίζαμε με τον πληθυσμό και όχι με, με την έκταση. Υπάρχουν θέματα όπως η ασφάλεια, Και όλα αυτά θα τα πούμε στην έκθεσή μας. Τώρα για την επίσκεψη στη Συρία, την αποστολή στη Συρία. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει διάλογος με όλους τους ενδιαφερομένους αν θέλουμε να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Να μιλήσουμε με όλους, αλλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μονομερώς αποφάσισαν να κόψουν τους διπλωματικούς δεσμούς με τη Συρία και από ό,τι ξέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το έχει πράξει με τους δεσμούς με, το, και με τη Βουλή της Συρίας δηλαδή. Επομένως ίσως το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ξαναρχίσουν οι επαφές είναι να ξανασυνδεθούμε με τη Συρία μέσω της Βουλής της. Έχουμε και την Εθνική Αντιπροσωπεία, συνεχίζουμε να μιλάμε και να συνομιλούμε με τη Συρία. Καλό θα ήταν ίσως τώρα αντί να μιλάμε περί αυτών να μιλάμε με αυτούς. Πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά στα σοβαρά και να δείξουμε ένα ελάχιστο όριο σεβασμού και αξιοπιστίας. Διάλογο δηλαδή με όλους τους ενδιαφερόμενους. Είναι και δικαίωμα και καθήκον μας να μπορούμε να συνομιλούμε με τους αντιστοίχους μας στην Συριακή κυβέρνηση. Αυτό ήθελα να σας τονίσω. Και με αυτή την ευκαιρία δεν ξέρω αν εσείς μιλάτε όλες τις γλώσσες εδώ στο Προεδρείο και αν τα καταλάβατε όλα όσα είπα, αλλά όσοι δεν βάλτε ακουστικά. Είναι καλό και σωστό να σέβεται κανείς τον ομιλητή. Είναι ντροπή να μας καλείτε εδώ για να σας πληροφορήσουμε για την αντιπροσωπεία αλλά να μην ακούτε καν τι λέμε. Δεν, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπαμε. Γιατί φαινόταν ότι δεν προσέχετε. Ενώ σε μια δημοκρατία πρέπει να τους ακούτε όλους αδιακρίτως και από τα πράγματα που σας αρέσουν και αυτά που δεν σας αρέσουν. Εγώ δεν θα τολμούσα να καλέσω κάποιον εδώ από την αντιπροσωπεία μας ρέκα ας πούμε να έρθει να μιλήσει και να μην τον ακούω. Μικρόφωνο Και επειδή σας άκουσα μπορώ και να σας απαντήσω τώρα. Εγώ ακούω πολύ. Αλλά θα μπορούσα να αναρωτηθώ και τι κάνατε στο ταξίδι. Αλλά δεν θα το πω τώρα. Τους τελευταίους 12-14 μήνες είχα πάει δύο φορές στο Λίβανο. στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Μία φορά μόνος μου και μία φορά με αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ. Και σε πιο... Ε, δεν μπορώ να σας ε, πω. Εκτός από τους Παλαιστινιακούς καταβλισμούς δεν έχουν φτιάξει άλλους καταβλισμού επίσημους, γιατί τους έχουν 60 χρόνια εκεί τους Παλαιστίνιους και έχουν ήδη πολλά προβλήματα με του καταβλισμού. Ε, και το γεγονός ότι σε μια χώρα που έχει κατοίκου 4 εκατομμύρια, οι πρόσφυγες είναι 1,3 περίπου, εκ των οποίων ε, ένα εκατομμύριο ίσως και παραπάνω από τον πόλεμο της Συρίας, δείχνει πόσο δραματική είναι η κατάσταση. Μια χώρα που είναι και ίδια θύμα πολέμων δι' αντιπροσώπων. Γιατί αυτό είναι το αποφασιστικό και θα ήθελα να το έχω ακούσει και στη δική σας έκθεση. Τι μπορούμε να κάνουμε στις συζητήσεις με το εκεί κοινοβούλιο για να φροντίσουμε να φέρουμε κοντά τις διάφορες ομάδες. 13-14 μήνες η χώρα είναι χωρίς πρόεδρο γιατί τα δύο χριστιανικά κόμματα δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους γιατί προβλέπεται από το Σύνταγμα να είναι χριστιανός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο περασμένο ταξίδι πριν από δύο μήνες είχαμε εντατικές διαβουλεύσεις με τα χριστιανικά κόμματα για να συμφωνήσουν επιτέλους σε ένα πρόσωπο για να αποκτήσει πρόεδρο η χώρα, πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είχαμε εντατικές συνομιλίες με ηθήνοντες, ηθήνοντες της Χεσπολά σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Και θα πρέπει να δούμε και να αναγνωρίσουμε ότι ένα χριστιανικό κόμμα και οι σύντες της Χεσπολά πώς να το πω, καθοδηγούνται και αναφέρουν στην Τεχεράνη, ενώ το Σουνητικό κόμμα που εκεί το δολοφονηθής πρώην Πρωθυπουργό Χαρίρη και το άλλο χριστιανικό κόμμα λογοδοτούν στο Ιράκ. Αυτά είναι ο Λίβανος. Είναι μια χώρα που δείχνει το σύνολο της τραγωδίας της περιοχής και τις ε, διαμάχες και τους πολέμους για το ποιος θα ηγηθεί στην περιοχή. Με ε, πυρήνες, Τεχεράνη και Ριάτ, αλλά όχι μόνο. Ε, ε υπάρχει και η Συρία. Μάλλον στο, ο ένας λογοδοτεί στην Τεχεράνη και όλος στο Ριάτ, όχι στο Ιράκ. Ε, έχουν γίνει λοιπόν εκεί πέρα πόλεμοι. Η Χεσμπολάχ συμμετείχε στον πόλεμο στη Συρία, το στρατιωτικό σχέλος των Λιβανέζων της Χεσμολάχ προς το Χαλέπι. Και προσπαθεί το ίσις να επεκταθεί και προς το Λίβανο. Εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν να σπάσουν αυτοί οι δεσμοί και να πούμε ποιες είναι οι ευθύνες του Ριάτ και της Τεχεράνης. Το είπαμε στο ταξίδι μας πριν από 15 μέρες και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και για το Λίβανο. Ε, βέβαια, ιδιαίτερα για το Ιράκ και για τη Σύρια. Πρέπει να σπάσουν, να κοπούν αυτά τα νήματα. Τώρα υπάρχει μια ευκαιρία, έχω την εντύπωση, με υπεύθυνη συμπεριφορά όλοι μας, να προχωρήσουμε. Και έχουμε ευθύνη όλοι που δημιουργήθηκε αυτό το έκτρωμα, το τέρας που λέγεται ίσης και δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει. Έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Αυτό το τέρας πρέπει να καταπολεμήσουμε. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει δυνατότητα με κοινοβουλευτική διαδικασία και αποστολή να πάμε στη Συρία. Είπατε να διαμεσολαβήσουμε αγαπητοί συνάδελφε. Εγώ δεν θα το τολμούσα. Εσείς πώς θέλετε ακριβώς να το κάνετε. Εγώ δεν θα το τολμούσα, δεν το αναλαμβάνω. Αν δούμε και την κυβέρνηση που θέλετε να έχετε επαφέ στη Συρία, αυτοί ρίχνουν βόβες βαρέλια σε άμαχο πληθυσμό στην ίδια τους χώρα, στον ίδιο τους το λαό. Τι γίνεται με τις χριστιανικές μειονότητες εκεί. Με τους ασυροχαλδαίους στο Ιράκ, τους Γεζιντή, άλλους Χαλδαίους στο Ιράκ και πολλούς άλλους. Όλες αυτές οι μειονότητες ζουν δράμα. Και τα κοινωνικά προβλήματα στο Λίβανο, που είναι σχετικά ευημερούσα χώρα, στην Ιορδανία είναι πολύ χειρότερα ως προς τις συνδίκες διαβίωσης λοιπά Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αν δεν λυθούν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα εκεί. Αυτό έχει σημασία και το λέω με κάθε ευγένεια. Πώς θα συνοδεύσουμε αυτό το μεγάλο γίγνεσθε εκεί, το πολιτικό. Στη Συρία, ας πούμε, αποτύχαμε. Διότι στην αρχική φάση της Συριακής κρίσης δεν είχαμε δυνατότητα να συζητήσουμε λογικά με τη Ρωσία που δεν θέλανε να βάλουν σε τάξη τον ε, Ασάντ. Αυτό είναι ένας παράγον. Και στο Ιράκ είναι η ανοησία του Αμερικανικού πολέμου. Πολλές βλακίες έχουν γίνει, αλλά θα πρέπει να το δούμε από κοινού ε, συνολικά και μόνο τότε θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε η Επιτροπή ΑΦΕΤ και την προσωπία που να πάει με έναν τρόπο παραγωγικό και χρήσιμο. Και σας ευχαριστώ που με ακούσατε και πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πείτε, Κυρία Ματίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω αυτά τα οποία λέτε. Ωστόσο, δεν αρκεί να εξετάζει κανείς τα πράγματα όντας εκτός με την απόσταση αυτή και να επιρρύπτει ευθύνε των ένα των άλλων και να επικρίνει κατά αυτόν τον τρόπο τι κάνουν οι μεν και τι κάνουν οι δε. Καλύτερα να δούμε εμεί τι μπορούμε να κάνουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Α δούμε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, α αξιολογήσουμε την ευθύνη αυτή και α ξεπεράσουμε λίγο, ας υπερβούμε πλέον απλώ τα ψηφίσματα, τι δηλώσεις, ας αναλάβουμε δράση επιτόπου. Ακόμα και αν αναλάβουμε δράση μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθούν κάποια πράγματα που ήδη τα γνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αυτός είναι ο ρόλος μας. Διαφορετικά για ποιο λόγο να υπάρχουν στη τελευταία ανάλυση και κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείε, για ποιο λόγο να, λόγο να εφίσταται η ίδια η Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουμε για να λάβουμε δράση εξ ονόματο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο Νομίζω ότι ε, θα ήταν πολύ περιορισμένο το έργο μας αν χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά του Ευρωπαίου Φερολογούμενου μόνο και μόνο για να συντάξουμε γνωμοδοτήσεις και ψηφίσματα, ενώ φαίνεται τελικά να αποφασίζουμε να μην αναλάβουμε επιτόπου δράση. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα πραγματικά δεν σας καταλαβαίνω. Εδώ η Επιτροπή μας και ο Πρόεδρος τη το τελευταίο 1,5 χρόνο μετέβησαν εκεί, σχεδόν σε όλους του καταβλισμούς των προσφύγων. Παρά τις προειδοποίησεις τότε, όταν έκλεισε το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, πήγαμε στη Βαγδάτη με τεράστιους κινδύνους που αναλάβαμε και ρίσκα. Με προσωπικές απειλές στις ε, περιοχές εκεί και να έρχεστε και να λέτε ότι δεν αρκεί αυτή η πολυθρόνα να τα κάνεις αυτά. Μήπως δεν ακούσατε τα πρώτα που σας είπα. Τώρα θα πρέπει να σταματήσουμε ε, ε, να ε, ξυβρίζουμε ο ένας τον άλλον για το ποιος είναι ο, ο, εκεί, δεν ξέρω, ο πιο αγωνιστής. Όλα αυτά τα συζητήσαμε, σας κάλεσα να παρευρεθείτε, να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας, τα πεπραγμένα της αντιπροσωπείας, μίλησαν και οι συνάδελφοι και καλά έγιναν. Τώρα αιτιάσεις και να ρίχνουμε ένας το φταίξιμο στον άλλον ποιος κάνει περισσότερα δεν γίνεται. Τουλάχιστον επειδή πήγατε τέσσερις μέρες στο Λίβανο δεν μπορείτε να παραγωνίστε τον πρόεδρο της Επιτροπής, κοιτάξτε τι έχετε κάνει εσείς, τι έχουμε κάνει εμείς και πώς πολιτικά μπορούμε να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το πιο λογικό νομίζω, παρά να εξηγούμε ένα στον άλλον τι γίνεται και να απευθύνουμε διάφορες αιτιάσεις και ποιος δουλεύει καλύτερα. Ευχαριστώ και τα μέλη της αντιπροσωπείας και σας είμαι ευγνώμων που αναλάβατε αυτό το βάρος της αντιπροσωπείας, κάνατε την παρουσίασή σας, τη συζητήσαμε. Έχω την άποψή μου και εγώ και την είπα για τα προβλήματα της περιοχής. Αυτό το τελευταίο που είπατε τώρα δεν το κατάλαβα. Και μην αρχίσουμε τώρα να βρίζουμε ένα στον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Eu peço Μα δεν ήθελα να επικρίνω κανέναν κύριε Πρόεδρε και πραγματικά ζητώ συγγνώμη. Απλώς είναι πολύ καλό να υπάρχει και η Επιτροπή, είναι πολύ καλό να υπάρχει και την προσωπία. Δεν αποδοκιμάζω κανέναν, δεν επικρίνω κανένα. Συμφωνώ με την τελευταία παρατηρήσή σας, ακριβώς όμω όπως η Επιτροπή σας κάνει τη δική σας τη δουλειά και εμείς κάνουμε τη δική μας. Η αντιπροσωπεία ανταποκρίνεται στην συγκεκριμένη εντολή που τη έχει δοθεί και θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό να υπάρχει μια επικοδομητική συνεργασία. Αυτό κάνουμε. Κάντε εσείς κάποιες συστάσεις, δεχτήκαμε τις συστάσεις και στη συνέχεια έκανα απλώς κάποιες παρατηρήσεις επί αυτών των συστάσεων. Μάλλον μιλάμε όμως για διαφορετικά πράγματα. Το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι σας ευχαριστώ προφανώς για την πρόσκλησή σας, για τη δυνατότητα που μας δώσετε να κάνουμε ένα απολογισμό της αποστολής μας και να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο για την αποστολή αυτή. Προφανώς θα πρέπει από κοινού να εργαστούμε, πρέπει να σημειώσουμε ακόμα πρόοδο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Ολοκληρώνω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτά τα τελευταία λόγια. Ίσως είμαι και εγώ πολύ ευαίσθητος και είναι γνωστό αυτό ότι είμαι μηγιάγκηχτος και αρπάχτηκα. Εντάξει, προχωρούμε και ελπίζω να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και ερχόμαστε τώρα στην επόμενη ανταλλαγή απόψε με την κυρία Μαγιορέγκο. Έχει φτάσει, είναι και κλεισμένο των θυρών.